Πίεση. Χθε, αγαπητοί συνάδελφοι, μια τρομοκρατική επίθεση έπληξε χθε την Τινησία, την πρωτεύουσα της Τινησίας. 14 μέλη της Προεδρικής φρουρά χάσαν τη ζωή τους. Εξ λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταδικάζω με τον πιο απόλυτο τρόπο αυτή την αποτρόπαια πράξη και θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τον τινησιακό λαό και την κυβέρνηση της Τινησίας. Εκφράζουμε επίσης αλληλεγγύη στις οικογένειες των θυμάτων. Μέσα σε δύο εβδομάδες χτύπησαν τρομοκράτες στη Βηρητό, το Παρίσι, τον Παμάκο και εκ νέου την ε, Τινησία και κάθε φορά προκαλούν ιδιαίτερο πόνο. Οι τρομοκράτες για μία ακόμη φορά όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όλοι μας Είμαστε δεσμευμένοι για το σημαντικό αυτό αγώνα που θα κρατήσει μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά θα διέπεται πάντα από φασιστικότητα και από τις δημοκρατικές μας αρχές και από μια ενισχυμένη συνεργασία με τους συμμάχους μας και τους εταίρους μας. Σας ευχαριστώ. Πρώτο λοιπόν σημείο τη ημερήσια διάταξη έχουμε τι δηλώσει του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής για τι τρομοκρατικέ επιθέσει στο Παρίσι. Και επ' αυτού έχει το λόγο ο Προεδρεύων του Συμβουλίου Σμιτ,